και Τι συνάδελφοι, αγαπητοί συνάδελφοι, κάντε ησυχία εκεί πέρα, Κομισιόν, Εξωτερική Υπηρεσία, σους. They follow you, Frederica, not me. Σένα, εσένα ακούνε, Φρεντερίκα, εμένα τίποτα. Ευχαριστώ πολύ που συμφωνήσετε να μας ενημερώσετε για την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας που αποφασίστηκε επισήμως στο Σώμα των Επιτρόπων σήμερα το πρωί. Καλωσορίζω την ύπατη εκπρόσωπο την κυρία Μογκερίνη και τον Επίτροπο τον κύριο Χάν. Νομίζω χρειαζόταν αυτό. Αλλά αν δει κανεί εξελίξεις ε, στα νότια και το τι έγινε στο Παρίσι που είχε κάποια σχέση οπωσδήποτε. Αν δούμε λοιπόν προς Ανατολάς όπου παρά τη συμφωνία του Μίνσκ δεν έχουμε κάποια ικανοποιητική λύση και την κατάσταση στη Μολδαβία και η Γεωργία που επίσης είναι ανησυχητική. Νομίζω πως πρέπει ε, έπρεπε να γίνει αυτή η συνάντηση για να μπορέσει και η Φεντερίκα να μας πει κάποια πράγματα για τη συνεδρία των Υπουργών Εξωτερικών τη Δευτέρα για να μπορέσουμε να το συζητήσουμε αυτό. Δεν θα κάνω εγώ κάποια εισαγωγή, αλλά θεωρώ πως πρέπει να γίνει μια συζήτηση ε, και μετά οι συντονιστές να έχουν δύο λεπτά ίσως 1,5 οι υπόλοιποι βουλευτές ένα λεπτό, ε, λεπτό. Και μία παρτέρα το πρέπει να ολοκληρώσουμε, άκουσα. Οπότε δεν υπάρχει πολύς χρόνος ούτως ή άλλως. Τέλος πάντων, θα συνεχιστεί η συζήτηση γιατί θα γράψουμε και εκθέσεις και τα σχετικά. τις επόμενες εβδομάδες. Οπότε δεν είναι η τελευταία συζήτηση, αλλά μια εισαγωγή στη συζήτηση. Γιατί μπορεί να επηρεάσει την μελλοντική μας πολιτική, ελπίζω δηλαδή. Κυρία, τι εκπρόσωπε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Έλμαρ. Σήμερα, μόλις τώρα στο Σώμα των Επιτρόπων, εγκρίναμε πρόταση για την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας. Αυτό ακολουθεί ενός έτους ευρύτατες διαβουλεύσεις με όλους τους ενδιαφερομένους από διάφορες προελεύσεις. Δεν εννοώ μόνο τις χώρες εταίρους, κυβερνήσεις, αλλά και κράτη-μέλη, ευρωπαϊκά ιδρύματα και θεσμούς, το Ευρωκοινοβούλιο το ίδιο, αλλά και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, τα εθνικά κοινοβούλια, τον επιχειρηματικό κόσμο, think tanks και πανεπιστήμια. Οι τόσο διαφορετικές απόψεις παρόλα αυτά συμφωνούν σε ένα σημείο να έχουμε ένα κοινό πλαίσιο για τους ε, εταίρους μας ε, στην ε, γεωγραφική ζώνη νότια και βόρεια μάλλον ανατολικά και νότια, αλλά όπως υπόθηκε, το πλαίσιο θα υπάρξει, θα είναι ένα, αλλά είναι σαφής και η ένδειξη ότι χρειάζεται αλλαγή. Αλλαγή στον τρόπο που ε, την πολιτική μας. Ένα νέο πρόσωπο και μια νέα αρχή για την πολιτική μας. Το σημερινό πολιτικό περιβάλλον, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά στην ευρύτερη περιοχή, φαίνεται ότι πρέπει να μεταβάλουμε τη στάση μας και τον τρόπο που ερμηνεύουμε την πολιτική γειτονίας. Όταν λέω πολιτική γειτονία, το λέω έτσι γιατί νομίζω ότι το πολιτικό σκηνικό, το, το σκηνικό ασφάλειας αυτό που βλέπουμε από τους εταίρους μας στην όλη περιοχή, αλλά και, ως, ε, και από τους Ευρωπαίους πολίτες στι περισσότερες περιπτώσει, βλέπουμε ότι πρέπει να περάσουμε από μια προσέγγιση που βασιζόταν την υπόθεση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο κέντρο και οι γείτονε γύρω μα που έρχονται λίγο πολύ προ το μέρο μα, πρέπει να περάσουμε σε μια θεώρηση που θα βασίζεται σε εταιρική σχέση ισότιμων εταίρων με παρόμοια προβλήματα, κάποιες φορές παρόμοιες ευκαιρίες και θα πρέπει να οικοδομήσουμε εργαλεία και πλατφόρμες επικοινωνίας για να συνεργαστούμε αποτελεσματικά και για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις, αλλά και για να δράξουμε τις ευκαιρίε. Θα πρέπει να δράξουμε ότι και οι προκλήσεις και οι ευκαιρίε που είναι κοινέ είναι διαφορετικές από ό,τι στο παρελθόν. Με τον Έλμαρ σκεφτήκαμε ότι θα μπορούσα να σα ενημερώσω λιγάκι και για το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών. Αυτό θα μπορούσε να γίνει με διαφορετικούς τρόπους, Ίσως δεν είναι εδώ η καλύτερη ευκαιρία να το κάνουμε, αλλά τη Δευτέρα με τους υπουργού Εξωτερικών και χθε με τους υπουργού Άμυνας προφανώς επικεντρωθήκαμε στις τρομοκρατικές επιθέσεις της Παρασκευής στο Παρίσι. Επίσης, στις επιθέσεις που προηγήθηκαν λίγες ώρες στη Βηρητό, και αυτές που πριν από λίγες εβδομάδες ε, στην Αίγυπτο έπληξαν το ρωσικό αεροπλάνο. Και γενικότερα στην Αίγυπτο, στο Ιράκ, στην Ισία ίσως να ήταν πάλι δράση του ίσως αυτό που είχε γίνει πριν από λίγους μήνες, βλέπουμε ότι στην ε, γεωγραφική μας ζώνη έχουμε τις ίδιες απειλές κατά της ασφαλείας μας. Γι' αυτό το είπα και χθε και το είπα και στον Γάλλο Υπουργό ε, Άμυνας, τον κύριο Λεντριά, ότι σκέψεις μας είναι στο Παρίσι για τις επιθέσεις αυτές, αλλά επίθεση δεν δέχτηκε μόνο όλη η Ευρώπη, αλλά οι κοινέ μας ρίζες, οι κοινέ μας πολιτιστικές αξίες. Σε αυτό αισθανόμαστε ότι δεχτήκαμε επίθεση όλοι. Και όλοι εδώ είμαστε ενωμένοι. Όπως και τους τελευταίους μήνες ανακαλύψαμε, κάποιοι από εμά από χρόνια, ότι η διαχείριση της κρίσης των μεταναστών και των προσφύγων μας αφορά όλους. Μας αφορούν λοιπόν όλους αυτά τα θέματα και από κοινού θα πρέπει να βρούμε μια λύση να δώσουμε τέλος στον πόλεμο της Συρίας όπως το περασμένο Σάββατο καθίσαμε γύρω από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων στη Βιέννη ε, και πριν από ένα δεκαπενθήμερο και ως ε, χώρες γειτονικές της Λιβύης θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ε, ζητήσουμε μια κυβέρνηση εθνικού, εθνικής σωτηρίας στη Λιβύη. Και στα Ανατολικά λοιπόν και στο Νότο έχουμε τι ίδιε απειλέ, ενδεχομένω και τι ίδιε ευκαιρίε και ήδη την περασμένη εβδομάδα όταν βρέθηκα στην Ουκρανία και τη Γεωργία ξέρω ότι ο επίτροπο Χάν θα πάει σήμερα και εκεί έχουμε κοινέ απειλέ κατά τη σταθερότητα καταρχάς, έπειτα και στατιωτικές πολλές φορές, απειλέ κατά της ενέργεια, κοινέ προκλήσει και ευκαιρίε λοιπόν και προ Συνολικά λοιπόν η ασφάλεια αλλά και το πολιτικό τοπίο γύρω από την Ευρώπη μας λένε ότι πρέπει να μετατυπιστούμε την προσέγγιση εταιρικής σχέσης. Πρέπει να αξιοποιήσουμε τα θεσμικά εργαλεία που έχουμε ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η νέα αρχή στις εταιρικές μας σχέσεις θα μπορέσει να μας επιτρέψει να οικοδομήσουμε σταθερά θεμέλια. Και αυτό αρκετά κατεπηγόντως. Ο επίτροπο Καν θα περάσει σε περισσότερε λεπτομέρειε για την αναθεωρημένη πολιτική αυτή καθεαυτή. Απλώς να αναφέρω πέντε αρχέ επί, επί των οποίων θα βασιστούμε. Και μάλιστα όλοι μαζί. Το τονίζω αυτό όλοι μαζί για τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι έχουμε συντονισμένη δράση και θέλω να ευχαριστήσω και τις υπηρεσίες μας που συνεργάστηκαν στενά μαζί μας όλη αυτή τη χρονιά και θα συνεχίσουν και μετά τη σημερινή ημέρα ώστε η εταιρική σχέση μας και η συνεργασία μας να συνεχιστούν και εκτός των Ευρωπαϊκών Θεσμικών κάνων. Ε, κάποιες αρχές για την πρόταση αυτή. Πρώτα απ' όλα να επικεντρωθούμε στην οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ιδίως για τις νέες γενιές. Αυτό αφορά και την Ευρώπη, δεν θα το συζητήσουμε αναγκαστικά μόνο στο επίπεδο αυτού του σχηματισμού κρατών μελών του Κοινοβουλίου, αλλά αφορά όλους τους νέους, όλη της Ευρώπης και της γειτονίας ε, και προς Ανατολάς και προς τον Νότο. Οικονομικές ευκαιρίες, δημιουργία θέσεων απασχόλησης και όχι μόνο ε, μέσα στην εκπαίδευση, αλλά δουλειέ για τους νέους και στα ανατολικά και στα νότια της Ευρωπαϊκής Πυρού. Αυτό είναι καθοριστική σημασία για τη σταθερότητα και την ειρηνική πορεία αυτών των χωρών και εντό τη Ευρώπη βέβαια. Ενεργειακή συνεργασία, δεύτερον, ε, ενέργεια. Έχουμε ενδείξει από όλου του ενδιαφερμένου ότι αυτό είναι ένα από τα θέματα, όχι μόνο προ Ανατολά αλλά και προ τον Νότο, που μπορούν να μα δώσουν έδαφο για να καλλιεργήσουμε μαζί κοινέ ευκαιρίε και κοινέ προκλήσει να αντιμετωπιστούν. Τρίτον, ασφάλεια. Γνωρίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονία δεν συμπεριλάμβανε εργαλεία για την ασφάλεια τώρα, δεν ήταν η πρώτη προτεραιότητα. Σήμερα όμω νομίζω καθίσταται σαφές ότι πρέπει να συμπεριλάβουμε ε, εργαλεία που μα δίνουν στα χέρια μα τα μέσα για να συνεργαστούμε με του εταίρου μα και προ Ανατολά και προ τον Νότο. Επίση, ανθεκτικότερε χώρε κοινωνίε και εξωτερικό και εσωτερικό για να μπορούν να αντιμετωπίσουν απειλέ. και ένα ευρύ φάσμα νέων πεδίων συνεργασία, λόγω χάρη με επικέντρωση στην πρόληψη των ε, συγκρούσεων και την μεταρρύθμιση του τομέα της ε, ασφάλειας. Πρέπει να, βρεθεί, να βρεθεί σωστή εξισορρόπηση μεταξύ τη αποδοτικότητα των μεταρρυθμίσεων στον τομέα της ασφάλειας και την ε, ε, ανοιχτή μορφή των κοινωνιών με, την, τον σεβασμό των βασικών αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέταρτο, προφανώς πάντοτε στο σκέλος της ασφάλειας τη όλη μα δουλειά, η αντιμετώπιση τη τρομοκρατία, τη ριζοσπαστικοποίηση, της χρηματοδότησης των δικτύων τρομοκρατών και η εντατική συνεργασία κατά του οργανωμένου εγκλήματος, της διαφθοράς, καθώς και οι διαφορετικές τάσεις ε, που πρέπει να αντιμετωπιστούν στον τομέα της ασφάλειας και να ληφθούν υπόψη. Και ε, επίσης η μετανάστευση, ε, νόμιμη και παράνομη, λαθρέα. Αυτά πρέπει να συμβαδίζουν. Και το τρίτο στοιχείο, ε, η προστασία των ε, προσφύγων. Εκεί συνεργαζόμαστε όλο και πιο στενά με του εταίρου μας και για τη δική τους και για τη δική μας, αλλά εδώ μας αφορά περισσότερο η δική μας πλευρά της ιστορίας, η δυνατότητα να ε, φιλοξενήσουμε, να υποδεχτούμε πρόσφυγες και να βεβαιωθούμε ότι λειτουργεί το σύστημα ασύλου και το σύστημα προστασία επαρκώ. Για την νόμιμη μετανάστευση, την θα πρέπει εδώ να στηρίξουμε την κινητικότητα, λαμβάνοντα υπόψη τι δημογραφικέ και οικονομικέ ανάγκε, ε, πρόθεσμα και μέσω μακρυπρόθεσμα, γιατί χρειαζόμαστε και την νόμιμη μετανάστευση, αλλά θα πρέπει να έχουμε και ανταλλαγέ φοιτητών, επιστημόνων, ερευνητών, επιχειρηματιών. Αυτή η κινητικότητα πρέπει να ενθαρρυνθεί, να βρούμε απλού τρόπου να διασυνδεθεί η Ευρώπη με τον υπόλοιπο κόσμο. Επίση, η παράτυπη μετανάστευση, η λαθρέα. Πρέπει να έχουμε μια κοινή διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Πρέπει να καταπολεμήσουμε του διακινητέ και του εμπόρου ανθρώπων και τι διασυνδέσει με άλλε εγκληματικέ ενδεχομένω οργανώσει, καθώ και κοινή εργασία για τι επιστροφέ και, τους... και τι επανεισδοχέ. Κοιτώντα τι μπορεί να είναι η επίδραση στι τοπικέ κοινότητε, με καλέ ευκαιρίε για τι τοπικέ κοινότητε ενδεχομένω. Πέμπτο και τελευταίο, θα πρέπει να ασχοληθούμε με το τι γίνεται στους γείτονες των γειτόνων μας. Δηλαδή, πέραν του αυστηρού γειτονικού περιβάλλοντος, θα πρέπει να ασχοληθούμε και με άλλους βασικούς εταίρους στον κόσμο για να δούμε τι κοινέ προκλήσεις μπορεί να έχουμε. Λόγω χάρη στην Αφρική, σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση, την ενέργεια, την ασφάλεια, την υγεία. Σκεφτείτε πόση δουλειά έχουμε κάνει για τον ιό έμπολα τελευταία μόλις χρονιά και φαίνεται τόσο μακρινό. Υπάρχουν λοιπόν διάβλοι που ανοίγουν μέσω των γειτόνων μας προς μακρινότερους γειτονές και τελικά καταλήγουν στην Ευρώπη ούτως ή άλλως. Θα ολοκληρώσω εδώ λέγοντας ότι ως προς τη διαδικασία, όπως είπε σήμερα, αυτή είναι μόλις η αρχή, όχι η αρχή γιατί αυτό το επεξεργαζόμαστε εδώ και ένα χρόνο μεν, αλλά ως προς την θεσμική μας συνεργασία δεν αυτό το τελευταίο κεφάλαιο, και μετά από αυτή την ανταλλαγή απόψεων με εσά, με το Κοινοβούλιο, θα συζητήσουμε την πρόταση με τα κάτι μέλη, με τις χώρες εταίρους, ξεχωριστά. Χθε συναντήσαμε τους πρέσβεις όλων των ενδιαφερομένων χωρών και θέλουμε να έχουμε διάλογο μεταξύ ισότιμων εταίρων. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε οι ποιότερες μεθόδους εργασίας. Είναι και αυτό μια πρόκληση, αλλά θα προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε τα γραφειοκρατική προσέγγιση που κάποιε φορέ έχουμε στι σχέσει με του συνεργάτε μα, το ίδιο και εκείνοι, οι εταίροι μα. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε μια πολιτικότερη, μια πιο πολιτική προσέγγιση και έναν αποτελεσματικότερο τρόπο να εξασφαλίσουμε και τη συμμετοχή τη κοινωνία των πολιτών παντού. Και προφανώ θα τηρούμε ενήμερο το Κοινοβούλιο, το Ευρωκοινοβούλιο, για να γνωρίζει το έργο μα. Äh, Πριν δώσω τον λόγο στον κύριο Χάν να υπενθυμίσω κάτι θα ήθελα να παρακαλέσω. Λόγω του αιτήματος γαλλικής κυβέρνησης ε, για το άρθρο 40... 42.7 να μας πει η ΣΕΝΤΕ τι μορφή θα μπορούσε να έχει ενεργοποιήσει αυτού του άρθρου πρακτικά. Καλό είναι λοιπόν να ετοιμάσετε ένα ενημερωτικό σημείωμα το τι σημαίνει αυτό πρακτικά. Εάν συμφωνείτε να θεωρώ ότι εγκρίνεται. Λοιπόν, ευχαριστώ. Τον λόγο έχει ο Γιωχάνες ε, Χάν. Ευχαριστώ Έλμα, για να συμπληρώσω την είπα τη εκπρόσωπο να πω το εξής ε, έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία επανεξέτασης της πολιτικής γειτονίας όχι γιατί θεωρούμε πως ε, όλα όσα έγιναν τα τελευταία δέκα χρόνια ήταν ε, λάθος αλλά γιατί λογικό είναι μετά από 10 χρόνια να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας ε, και με βάση την ε, τρέχουσα κατάσταση για να δούμε πώς θεωρούμε ότι θα πρέπει να διαμορφωθεί η σχέση με τις γειτονικέ μας χώρες τα επόμενα 10 χρόνια. Οπότε το έγγραφο αυτό μπορεί να θεωρηθεί ένα είδος κατευθυντηρίων γραμμών για το πώς θα μπορέσουμε να διαμορφώσουμε τη σχέση μας με τους γειτονές μας. Λοιπόν, θα πρέπει όσον αφορά την νότια γειτονία να επιδείξουμε εντονότερα το ενδιαφέρον μας για να κατοχυρώσουμε και τα συμφέροντά μας. Γιατί ήμασταν κάπως πολύ ευγενικοί και επιφυλακτικοί γιατί ενώ τα συμφέροντα μας είναι κοινά με τους γείτονες, δηλαδή η ειρήνη, η σταθερότητα και η ευημερία, και αν υπάρχουν αυτά, εποφελούμαστε και εμείς στην Ευρώπη. Σκεφτείτε την τωρινή μεταναστευτική πίεση. Δεν θα υπήρχε αν υπήρχε σε αυτές τις χώρες ε, ευημερία και σταθερότητα. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ποια είναι η δουλειά μας τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή να διασφαλίσουμε πως ε, θα υπάρχει σταθερότητα, να σταθεροποιηθεί η κατάσταση στις γειτονικές μας ε, χώρες, γιατί όπως ε, γνωρίζετε έχουμε πάνω από 20 εκατομμύρια πρόσφυγες και εκτοπισμένους στις γειτονικές μας χώρες. Έχουμε πάνω από 10 ενοπλές συγκρούσεις στη γειτονιά μας. Έχουμε και εξελίξεις ε, στο θέμα του κράτους ε, δικαίου όπου έχουμε μια επιδίνωση ή τουλάχιστον δεν υπάρχει βελτίωση. Οπότε λογικό είναι νομίζω να ορίσουμε τα βασικά σημεία αυτής της πολιτικής τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές εδώ μέσα, οπότε η διαδικασία αυτή της ε, διαβούλευσης έχει εμπλέξει πάρα πολλές χώρες, οργανώσεις, ε, ΜΚΟ και ιδιώτες και ακριβώς επιβεβαιώνει αυτό το οποίο ε, γράψαμε και στο σχέδιο ότι δηλαδή θα πρέπει πρώτα απ' όλα να έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση για την κάθε χώρα ξεχωριστά. Δεύτερον, να υπάρξει μια θεματική εστίαση, η Φεντερίκα Μοργκερίνη το ανέφερε ήδη, κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει μέχρι το τέλος της ε, εντολής μας. Ένα τέτοιο θέμα παραδείγματο χάρη είναι η ενέργεια και όλα αυτά τα οποία καλύπτονται από το λεγόμενο people to people, ειδικά η επαφή με την νεολαία και οπωσδήποτε ως μια ευρύτερη διάσταση η οικονομική ανάπτυξη. Δεύτερον, είναι σημαντικό να τα αγκαλιάσουν αυτά και οι εταίροι μας. Δεν πρέπει αυτά να θεωρηθούν ένας μονόδρομος, αλλά μια λεωφόρος διπλής κατεύθυνσης, στην οποία θα συναντηθούμε. Αναφέρθηκαν ήδη το ότι θα πρέπει, αναφέρθηκα στο ότι θα πρέπει να συζητάμε τα θέματα που αφορούν την κάθε χώρα ξεχωριστά. Δεν μιλάμε με όλους για όλα, αλλά θα ασχοληθούμε με αυτά τα οποία μας απασχολούν. Και οπωσδήποτε θα πρέπει να έχουμε έναν πιο μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα και να αναπτύξουμε μία κάποια ευελιξία θα ήθελα επίσης να ξεκαθαρίσω πως θα πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ των κονδυλίων Ανατολικής και Νότιας Γειτονίας που έχει μία αναλογία 2 προς 1 και δεν πρέπει να αλλάξει. Αλλά στο εσωτερικό αυτών των δύο φακέλων χρειάζεται περισσότερη ευελιξία. Οπωσδήποτε Μπορεί κάποια στιγμή να υπάρξει μια εξισορρόπηση, αλλά απλούστατα αυτή τη στιγμή χρειάζεται να επενδύσουμε μαζικά στο Λίβανο και στην Ιορδανία για να στηρίξουμε αυτές τις χώρες για να αντιμετωπίσουν ακριβώς ε, τις προσφυγικές ροές. Από την άλλη έχουμε μια κατάσταση όπου θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα βήματα που πρέπει να κάνουμε και να παρέμβουμε εάν απαιτούνται κάποιες ε, περαιτέρω δράσεις. Τώρα, κάτι άλλο το οποίο προέκυψε κατά τη διάρκεια των ε, διαβουλεύσεων ήταν ακριβώς το ότι πέρα από τις διμερείς ε, σχέσεις πρέπει να δούμε και την συνεργασία σε ένα υπερεθνικό επίπεδο π.χ. τις χώρες του Μαγκρέμπ ή τον Νότιο Κάφκασο υπάρχει νομίζω εδώ πέρα υπάρχουν πολλές δυνατότητες και αν μιλάμε για σταθεροποίηση και τα λοιπά θα πρέπει ακριβώς να φροντίσουμε οι χώρες αυτές να αναπτύξουν σχέσεις μεταξύ τους όχι μόνο πολεμικές ε, συγκρούσεις αλλά να υπάρχει και κάποια ειρηνική ανταλλαγή απόψεων και θεωρώ πως ε, σημαντικό ε, είναι όσον αφορά την Μεσόγειο να δούμε τις δυνατότητες της Ένωσης για την Μεσόγειο Βεβαίω εδώ πέρα ο κάθε υπουργό έχει και το κάθε υπουργείο έχει ένα δικό του τρόπο που οργανώνει τις ε, συναντήσεις. Και ακριβώς ε, βεβαίως υπάρχει η διαδικασία της Βαρκελόνης ε, και Νομίζω πως ε, και από τη Ρίγα βγήκε ενισχυμένη η Ένωση για τη Μεσόγειο. Οπότε ήδη έχουμε ε, υπογράψει η Φεντερίκα Μοργκερίνη και η ταπεινότης μου και όλοι οι Υπουργοί Εξωτερικών των γειτονικών χωρών έχουμε δεσμευτεί σε αυτό το έγγραφο για να δούμε ακριβώς το ποιες είναι οι δυνατότητες που μπορούμε να έχουμε. Για να δούμε ακριβώς ε, το τι θα γίνει. Για να δούμε αν χρειάζεται και όταν χρειάζεται κάποια αναφορά να γράφουμε κάποια αναφορά. Δεν χρειάζεται να γίνεται αυτό μονίμως, εκθέσεις και εκθέσεις, αν δεν υπάρχει λόγος. Και τέλος, θα ήθελα να αφαιρθώ σε ένα πράγμα συγκεκριμένο. Αν έχουμε μια ρεαλιστική προσέγγιση, αυτό βεβαίως δεν είναι εις βάρος των θεμελιωδών μεγεθών είναι ξεκάθαρο νομίζω αυτό και αδιαπραγμάτευτο. Αλλά το ζήτημα είναι πώς θα διαφυλάξουμε τις βασικές αρχές για τις οποίες θεωρούμε πως πρέπει ε, να μπορεί να αναπτυχθεί μια κοινωνία ελεύθερη και με ευημερία πώς ακριβώς ε, θα εφαρμοστούν ε, στην κάθε χώρα στη μορφή που πρέπει χωρίς μετά αυτές οι χώρες ε, να βρεθούν σε κάποια δυσκολία. Στόχος μας πρέπει να είναι να αναπτύξουμε τα πράγματα έτσι ώστε οι αρχές του κράτους δικαίου, της αηφορίας να εφαρμοστούν και να υπάρχει ελευθερία των ΜΜΕ, του συνέρχεστε, ανεξαρτησία της δικαιοσύνη, όλα αυτά. Και αυτό θα γίνει με μια ενεργή πολιτική γειτονία. Σας ευχαριστώ. Herzlichen Dank. Wir haben eine gute halbe Stunde. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε μισή ώρα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ε, 22 άτομα έχουν ζητήσει το λόγο. Γι' αυτό παρακαλώ οι συντονιστές να μιλήσουν 1,5 λεπτό, οι υπόλοιποι ακόμη λιγότερο. Τον λόγο έχει ο κύριος Πρέντα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την ύπατη εκπρόσωπο και τον Επίτροπο Χαν για τις παρουσιάσεις τους. Θέλω να χαιρετήσω τις προτάσεις που υιοθετήθηκαν σήμερα και που θα εξετάσουμε σε βάθος. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ξέρουμε τι έχουμε κάνει σε σχέση με τις προσδοκίες που είχαμε εκφράσει με την έκθεση Κούκαν πριν από μερικούς μήνες. Ήδη από τότε μιλούσαμε για την πολιτική γειτονία που να βασίζεται στην πρόθεση αξιών, λαμβάνοντα υπόψη του πλαισίου ε, για την κάθε χώρα χωριστά και με ευελιξία για να εφαρμόζεται όσο γίνεται καλύτερα στην περίπτωση της κάθε χώρας. Χαίρομαι λοιπόν που βλέπω ότι η σταθεροποίηση εντοπίζεται ως η πιο σημαντική πρόκληση το πραγματικό διακύβευμα είναι ακριβώς αυτό, πώς θα έχουμε τα σταθερότητα μέσα στην πολυμορφία. Θέλω να στηρίξω επίσης και αυτό που ζήτησε ο πρόεδρός μας, ο κύριος Μπροκ. Είχαμε ανταλλαγή υπόψεων με τον κύριο Στάνι μέχρι τη Δευτέρα και συζητήσαμε για τη δυνατότητα κάποιας δράσης βάσει του άρθρου 222. Τώρα βλέπουμε ότι είναι η αμοιβαία άμυνα, το άρθρο αυτό το οποίο ενεργοποιείται γιατί πρόκειται για στρατιωτικές επιθέσεις. Έχει να κάνει με στρατιωτικές επιθέσεις, οπότε δεν είναι μόνο η τρομοκρατία. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας ε, πράγματι και σας ευχαριστώ. Να ξέρουμε τι περιλαμβάνει ακριβώς αυτή η δράση μας. Πρόεδρε, είπατε η Επίτροπε Επιτρέψτε μου να σας ε, ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Και θέλω επίσης να ευχαριστήσω και τον συγκεκριτή τον κύριο Κούκαν για την αξιόλογη δουλειά του. Κυρίως για την αναθεώρηση όσον αφορά του σοσιαλιστές θα μιλήσω και για την και εκ μέλους αντιπροσωπείας για τη Μολδαβία. Το θέμα του προσφυγικού και η τραγωδία αυτή των, που ζουν οι πρόσφυγες είναι άνευ προηγουμένου και απαιτεί την αρρωγή μας, τη βοήθειά μας και την αμεσοδράση μας. Όμως, σας κάνω έκκληση, δεδομένου ότι το πρόβλημα συνεχίζεται και θα καταλήξουμε σε ένα δίλημα ανατολικά ή νότια να βοηθήσουμε, πρέπει να έχουμε μια σφαιρική άποψη. Το Κοινοβούλιο κατάφερε να πετύχει σύγκληση με ένα φιλόδοξο κείμενο και αν δούμε το έγγραφο που μας δώσατε και ακούγοντά σας, βλέπω πολλές κοινέ απειλές στις ε, συζητήσεις και στα πράγματα που φασίστε να αντιμετωπίσετε. Η ερώτηση μου είναι η Η αναθεώρηση περιλαμβάνει και κάποιες φιλόδοξες πρωτοβουλίες που συνοδεύονται από νέα μέσα. Πώς προβλέπετε τη χρηματοδότησή τους. Θα υπάρξουν νέοι πόροι ή θα υπάρξει ανακατανομή των ε, πόρων που ήδη υπάρχουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε. Ευχαριστούμε για την ε, προσέλευσή σας και για, για την παρουσίαση από τον Επίτροπο. Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονία θα έπρεπε να συμβάλλει στην οικοδόμηση ενός ασφαλέστερου κόσμου για τις χώρες μας. Θα πρέπει λοιπόν να στηρίξουμε διαδικασίες επανοικοδόμησης της κοινωνίας των πολιτών, της ζωής των πολιτών στην Ευρώπη, στο νότο της Ευρώπης και χώρες όπως η Ουκρανία και η Γεωργία, αλλά κυρίως η Γεωργία. Ε, η Ουκρανία ας πούμε ότι είναι διαφορετική περίπτωση και έχει τα δικά της προβλήματα ασφάλειας. Όμως, ένα από τα σοβαρότερα ζητήματα είναι αυτό της παράνομης μετανάστευσης από τον Νότο. Γι' αυτό θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε τον διάλογο που συνοδεύει την πολιτική γειτονία, διότι χρειάζεται η συνεργασία με τους εταίρους μας, πρέπει να είναι αρκετά συγκεκριμένη και γι' αυτό θα πρέπει να δούμε τι, δραστηριότητα, τι δράση θα αναπτύξουμε στο μέλλον ώστε στις χώρες της νότιας όχθης της Μεσογείου να υπάρχει περισσότερη δραστηριοποίηση για την καταπολέμηση των δικτύων εμπόρων ε, ανθρώπων, των ε, δικτύων λαθρομετανάστευσης και τα μέτρα που πρέπει το Συμβούλιο πριν από έξι μήνες και δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί, υλοποιηθεί επιτέλου να γίνει πράξη. Ε, κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Μιλάμε για τη συνεργασία των χωρών ε, στη νότια αυτή τη Μεσογείου, αλλά δείτε τι γίνεται και στην Τουρκία. Μόνο περιθωριακά δείχτηκε το θέμα της ε, συνεργασίας για την καταπολέμηση αυτής της μαθίας, αυτού του παράνομου δικτύου. Ας σκεφτούμε λιγάκι μακροπρόθεσμα, σε έναν ορίζοντα πιο μακροπρόθεσμο. Να σκεφτούμε για τις πιο κοντινές απειλές αυτές τις μεταναστευτικές ροές που μετακινούνται προς την ε, Μαύρη Θάλασσα, τον Εύξηνο Πόντο. Οι διακινητές δραστηριοποιούνται στην Τουρκία στο νότο της Τουρκίας, όμως θα μπορούσαν να μετατοπιστούν και προς, την, ε, προς τον πόντω. πόντο. Ας αναρωτηθούμε λοιπόν πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τα μέτρα μας για να δώσουμε τέρμα και σε όλα αυτά. Μίλησατε πάρα πολύ, τέλος πάντων ο κύριος Αστροβίτσιος. Ευχαριστώ. Είπατε εκπρόσωπε, κύριε Επίτροπε. Ένα λεπτό. Α, όχι, είσαστε συντονιστής. Εντάξει, ένα μισή λεπτό έχετε τότε. Εντάξει, πρόεδρε, ναι, κάνετε διακρίσει κατά των φιλελεύθερων πάντα, είναι γνωστό. Με χαρά, λέει ο κύριος Μπροκ. Καλή αρχή. Συνεχίζει ο κύριος Αστρόβιτης. Τις τελευταίες δεκαετίες η πολιτική γειτονία είναι μέρος της ε, γενικότερης ευρωπαϊκής πολιτικής και για την ασφάλεια και για την ανάπτυξη και για την αλληλεγγύη. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει παρεξήγηση πάνω σε αυτό. Και στην πραγματικότητα θα έπρεπε να δούμε την ευρωπαϊκή γειτονία ως μια ευκαιρία και όχι ως ένα κίνδυνο για να έχουμε ένα περισσότερο ασφαλές μέλλον. Εκτιμάω ιδιαίτερα την έκθεση που μας παρουσιάσατε. Είναι πρακτική, λογική, ρεαλιστική και διαφορετικό το έγγραφο αυτό από τα προηγούμενα αντίστοιχα έγγραφα που είχαμε για την ευρωπαϊκή γειτονία. Είναι καλό που μπόρεσε να δει το φως στο έγγραφο αυτό. Εκτιμώ όλους ιδιαίτερος τόσα λέτε για την προβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πράγματι, επιτέλους το καταλάβαμε, γιατί δεν είναι δυνατόν να μένουμε στη σκιά τη στιγμή που προσφέρουμε και κάνουμε πράγματα. Δύο σημεία θέλω να σας ρωτήσω να μου εξηγήσετε. Για τη συνεργασία και πά. Έχετε υπόψη σας κάτι ώστε άμεσα να δράσουμε. Θα έπρεπε. Δεύτερον, οι αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής πολιτικής επιτόπου. Προβλέπεται περισσότερη οικονομική στήριξη, περισσότερο προσωπικό στις αντιπροσωπείες μας στις χώρες που βρίσκονται στα πλαίσια της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας. Ευχαριστώ. Το πρώτο ερώτημά μου αφορά τη Συρία. Ποιες ε, πιθανότητες και βήματα βλέπετε κυρία Μογκερίνη να έρθει σε επαφή η κυβέρνηση με την αντιπολίτευση και τι μπορεί να γίνει για να μιλήσουμε με τις αντιπολιτευτικές ομάδες. Επίσης, ε, ποια είναι η εκτίμησή σας γιατί ο Ασάντ, ε, ε, για το αν ο Ασάντ είναι διατεθειμένος να προχωρήσει σε εκλογές. Επίσης, μιλάτε για πιο εύρωστες χώρες. Για ποιους τομείς μιλάτε Ποιου τομεί έχετε κατά νου, μιλάτε για πιο εύρωστες κοινωνίες, ε, κάτι είπε και ο κύριο Χάν ανάλογο. Μετά, οι κοινωνίες οι εύρωστες είναι οι δικαιότερε ε, κοινωνίες ε, που περιλαμβάνουν όλες τις ομάδες, όπως παραδείγματο χάρη του Σουνίτε του Ιράκ. Τι μέτρα θα μπορούσαν να ληφθούν. Μιλήσαμε για επικίνδυνες ε, διάβλους. Οι πιο επικίνδυνες διάβλοι αυτή τη στιγμή είναι αυτοί που στηρίζουν το Ισλαμικό κράτος. Υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα για να σταματήσει η οικονομική στήριξη και η στήριξη στον τομέα της επιμελητίας και του εφοδιασμού στο επίπεδο του οπλισμού. Π.χ. σκοπεύετε να κάνετε κάτι σε σχέση με το Κατάρ. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Μην ξεχνάμε ότι το θέμα είναι η μεταρρύθμιση της ε, πολιτικής γειτονίας. Δεν είναι εδώ πέρα η συζήτηση για τη, για τη Συρία και τη διαδικασία της γέννης. Αυτή θα γίνει, θα συνεχιστεί και τη Δευτέρα κτλ. Λοιπόν, Χάουταλα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε. Μια καλή συνεργασία μεταξύ σας οδήγησε στο να, στο να εντοπίσουμε νέους τομείς για συνεργασία, για παράδειγμα στο τομέα της ασφάλειας. Και βέβαια και συμφωνώ απόλυτα με τον Επίτροπο Χάν που είπε ότι η φτώχεια, η διαφθορά και η κακή διακυβέρνηση αποτελούν πηγές ανασφάλειας. Και ακριβώς έτσι βλέπουμε που είναι οι προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε για να πετύχουμε τη σταθερότητα. Πρέπει όπως προτείνετε κι εσείς να μείνουμε στα θεμελιώδη, όπως τα είπατε, κύριε Χάν, την μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, ανεξαρτησία του συστήματος αυτού και καπολέμηση της διαφθοράς. Σίγουρα τέτοιες εξελίξεις θέλουμε να δούμε, όπως και οικονομικές ευκαιρίες σε αυτές τις χώρες. Τώρα, για την διάσταση της ασφάλειας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πράγματι υπάρχουν πάρα πολλές ε, διενέξεις στην περιοχή και ανατολικά και νότια της Ευρώπης. Άρα την πρόληψη και την επίλυση ακόμα και των παγωμένων διενέξεων που έχουμε σε πολλές από αυτές τις περιοχές. Εσείς λέτε η αρχή περισσότερα για περισσότερα θα, παραμείνει, αλλά ότι δεν φτάνει για να γίνουν οι μεταρρυθμίσεις που θα έπρεπε να γίνουν σε χώρες που ήδη έχουν δεσμευτεί. Στην πράξη όμως τι σημαίνει αυτό. Και έπειτα, εσείς αναφερθήκατε στους γείτονες των γειτόνων μας. Μιλήσατε για κοινοβουλευτική συνεργασία, Euronest, ε, σχέσεις με τα κοινοβούλια λοιπόν των χωρών αυτών που είναι γείτονες των γειτόνων μας. Τι λέτε γι' αυτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. με την πρόσκληση να παραμένουμε εντός θέματος Εκμεταλλεύομαι την ευκαιρία για να πω ότι αυτά τα τα γεγονότα πρέπει να μα ανοίξουν τα μάτια. Και η πολιτική γειτονία πρέπει να αναθεωρηθεί υπό το φω των όσων συμβαίνουν που αλλάζουν τελείω τι ισορροπίε στην Ευρώπη. Την πολιτική τη γειτονία πώ θα την αναθεωρήσουμε χωρί να λαμβάνουμε υπόψη το γεγονό ότι έρχονται πρόσφυγε οι οποίοι ενδεχομένω να είναι συνδεδεμένοι και να έχουν σχέση με το ΙΖΙΣ. Επίσης, οι χώρες ε, γειτονικέ και οι γείτονες των γειτόνων μας θα μπορούσαν να βρίσκονται στον κατάλογο των 40 χωρών που χρηματοδοτούν το ΙΖΙΣ. Με, μέσω της Τουρκίας πηγαίνουν χρηματοδοτήσεις ε, και τη λαθρέα πώληση πετρελαίου, χρήματα και ποσά στα χέρια των τρομοκρατών του ΙΖΙΣ. Εκεί πρέπει να επικεντρωθεί η συζήτησή μας. Εδώ, στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, όμως συνέβησαν στο Παρίσι και τις Βρυξέλλες. Το να μην συζητάμε για αυτά είναι τελείω εκτός πραγματικότητα. Mr. Chairman. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλωσορίζω την παρουσίαση της αναθεώρησης πολιτικής γειτονίας από τους ε, έξοχους καλεσμένους μας. Είναι ζωτική σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις σχέσεις με τους εταίρους της στην γεωγραφική αυτή ζώνη να πάρει η πολιτική την σωστή πορεία. Αγωνιζόμαστε σε μια περίοδο κρίσης και προκλήσεων στην πολύ κοντινή γειτονιά μας και που επηρεάζει με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, ε, ορατό πλέον, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην έκθεση μου αναφέρθηκα στην επιστροφή στις βασικές ε, αρχές, δηλαδή να ε, έχουμε περισσότερη εμπλοκή σε θεμελιώδους σημασία ζητήματα. Αυτό καλώς το λαμβάνει υπόψη η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονία, καθώς και πολλά άλλα στοιχεία. Ερχόμενοι αντιμέτωπο με τις πρόσφατες αλλά και τις επερχόμενες προκλήσεις, θα πρέπει να αντιδρούμε εγκαίρως. Αυτό ήταν ε, από πολύ καιρό ένα πρόβλημα. Γι' αυτό τώρα περισσότερο από ποτέ θα πρέπει να έχουμε μια πολιτική κοινωνία που να βασίζεται περισσότερο σε πολιτικέ προτεραιότητε και θα καλέσω και του δύο εξαιρετού καλεσμένου μα να δείξουν περισσότερο έντονη παρουσία στην όλη περιοχή σε ό,τι αφορά τι πολιτικέ μα δράσει. Δεν μπορούμε να συνεχίζουμε σε να μην έχει αλλάξει τίποτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία η παρουσίαση, όμως πάντοτε ανησυχώ. Γιατί όταν έχουμε τέτοια σοβαρά γεγονότα πρέπει να διατηρούμε και την κοινή μας λογική. Και πολλά από αυτά που μπορούμε να γράψουμε σε ένα κείμενο είναι πολύ διαφορετικό. Η ισορροπία μεταξύ δικαίου και ελευθερίας, σταθερότητα και ελευθερίας. Θα πρέπει να δούμε στρατηγικώς τι έχει αλλάξει στην περιοχή μας σε σχέση με το παρελθόν αλλά υπάρχουν και κάποιε ερωτήσει που ε, δεν έχουμε απαντήσει ω σήμερα. Διαφεύγουμε διαρκώ. Πώ μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεσματικά να προωθήσει την κοινωνική σταθερότητα σε ε, στα περιβάλλοντα. Αυτό είναι ένα θέμα. Επίση, πώ να συνεργαστεί με του τοπικού ε, περιφερειακού φορεί αλλά και του διεθνεί πρωταγωνιστέ για την προώθηση τη ειρήνη. Και τέλο, τι σχέση μπορεί να υπάρχει μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονία όσα λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, πέραν των απλών λόγων. Διότι τέτοια συζήτηση δεν γίνεται. Η νέα ισορροπία που πρέπει να εξεύρουμε στι συμφωνίε ελευθερών συναλλαγών και την πολιτική συνεργασία. Αυτά είναι ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε διαρκώ. Και ε, υπό αυτό το φω θα πρέπει να δούμε και το θέμα τη μετανάστευση. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα για το ότι έχουμε αυτό το έγγραφο, το οποίο είναι αναλωτικό, έχει αρκετό όραμα θα έλεγα, αλλά εγώ θα περίμενα επίδειξη περισσότερης ηγεσία από τους Ευρωπαίους ηγέτες. Αυτό το οποίο λείπει και θα ήθελα να εστιάσω εδώ πέρα στις μεθόδους εργασίας Ε, κοιτάξτε, όταν μιλάμε για εξωτερική πολιτική και διπλωματία πρέπει να δρούμε εκεί όπου η κατάσταση είναι κρίσιμη, όπου υπάρχουν προβλήματα και προβλήματα που ξέρουμε επί σειρά ετών. Θα ήθελα λοιπόν κυρία Μογκερίνη να σας ζητήσω να εργαστείτε σε συγκεκριμένα προγράμματα δράσης για τις γνωστές ε, καταστάσεις ε, που έχουμε. Η κρίση που αύριο μπορεί να εξελιχθεί σε πολύ ε, επικίνδυνη κατεύθυνση. Τελείωσε ο χρόνος σας λέει ο πρόεδρος. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και για τις ε, προτάσεις σας ε, και συμφωνώ κυρία Μογκερίνη, κύριε Χάν όταν λέτε πως χρειαζόμαστε νέα κατεύθυνση της πολιτικής ε, γειτονίας και να στραφούμε στις χώρες αυτές της γειτονίας. Δηλαδή τι λέω, τι εννοώ, αν τα πάνε καλά οι γειτονέ μα, θα πηγαίνουν και για μας καλά τα πράγματα. Πρέπει να δούμε λοιπόν πώ αλλάξουν οι κοινωνικέ σχέσεις σε αυτές τις χώρε. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε ακριβώ ποιε θα είναι οι προτεραιότητες για την οικονομική ανάπτυξη και τη σταθερότητα. Ποια αποτελεσματικά νέα μέσα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε προς Νότον και προς Ανατολάς γιατί έχουμε τη δική μας την ανεργία των νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει ταυτόχρονα να σκεφτούμε τι θα κάνουμε και για αυτές τις χώρες και γενικά πώς θα καταπολεμήσουμε την ανεργία. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Ευχαριστώ. Thank you. I would also like... Η κυρία Λούνατσεκ, ευχαριστώ και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτά τα οποία μας είπατε και υπήρχε πράγματι τα τελευταία χρόνια πρόοδος στις σχέσεις ε, Γειτονία ε, και προς Ανατολάς και προς Νότον και τα εξηγήσατε αυτά. Ε, δηλαδή κάποια πράγματα πρέπει να τα δούμε πλέον ε, διαφορετικά και όπως είπε και συνάδελφος ο κ. Χάουταλα αναφέρατε και οι δύο σε ζητήματα εκτός του πλαισίου ασφαλείας. αναφέρατε την αδικία, φτώχεια, ανισότητα, διαφθορά και αυτό το οποίο ε, δεν βλέπω, δεν βλέπω στο κείμενο, το είπατε, είναι η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα και το συγκεκριμένο μου ερώτημα αφορά ακριβώς το ζήτημα του more for more που λέμε και χρειαζόμαστε κάποια αποτελεσματικότερη εμπλοκή. Ε, αυτό όμως θα πρέπει να σημαίνει less for less, δηλαδή αν μειωθεί η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα να δίνουμε και λιγότερα. Ε, η σταθερότητα χρειάζεται και δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα. Και ένα άλλο ερώτημα για την Ιεμένη. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, ο χρόνος σας τελείωσε, λέει ο Τι θα κάνετε για τη Σαουδική Αραβία, είπε η κυρία Λουνατσέκ. Ο κύριος Πλένκοβιτς. Και παρακαλώ να είστε ευγενείς με τους συναδέλφους, κύριε Πλένκοβιτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστούμε κυρία Μογκερίνη, Επίτροπε Χάνη. Νομίζω ότι το έγγραφο που μα παρουσιάζεται είναι πραγματικά πολύ έγκυρο. Και τόση προετοιμασία με την εξωτερική πολιτική, τους στόχους αναπτυξιακής πολιτικής. Νομίζω έχουμε πυλώνες εξωτερικής πολιτικής σημαντικούς για την Επιτροπή μας και με δουλειά ετών πίσω. Είναι πολύ, κάτι που εκτιμούμε πολύ λοιπόν. Ε, ήθελα να ρωτήσω στην προσπάθεια να ενισχύσουμε κάποια κράτη πώς θα εκμεταλλευτείτε τις συμφωνίες σύνδεσης. Είναι δύο σημεία κλειδί που άκουσα από την αναφορά σας σήμερα ε, για την σταθεροποίηση και την εταιρική σχέση. Πώ θα τα αξιοποιήσετε στην εξωτερική μα πολιτική και επίση στα δημοσιονομικά μα μέσα. Το Κοινοβούλιο στέλνει πολύ σαφεί ενδείξει για την κρίση των μεταναστών, για τι δράσει εξωτερική πολιτική και το τι θα πρέπει να γίνει στον προπολογισμό του 2016. Και επίση η καλύτερη χρήση των πολυμερών ε, φόρα που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν καλύτερα για να υπάρχει συζήτηση για συγκεκριμένα προβλήματα στην γεωγραφική αυτή ζώνη. Ευχαριστούμε κυρία Βαλεντιάνο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Μογκερίνη, κύριε Χάν, σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε να μας παρουσιάσετε τη δουλειά αυτή που είναι σε βάθος και σοβαρή. Θέλω να ρωτήσω κάτι για μας τους ίδιους. Δηλαδή, χρειαζόμαστε σταθερούς γείτονες. Ναι. Η συμπεριφορά όμως κάποιων χωρών μελών έχει σαν αποτέλεσμα να μην μπορεί να το πετύχει αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν ε, η Ουγγαρία πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο την απόφαση για την κατανομή των προσφύγων και η Σλοβακία κάνει τα δικά της, τότε πώς εμείς θα έχουμε αξιοπιστία για να πετύχουμε τη συνεργασία και τη σταθερότητα με τους γειτονές μας. Πώς θα τα πηγαίνουμε καλά με τους γειτονές μας αν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Πώς θα πειράσουμε τον περιγυρό μας. Λοιπόν, μην κοιτάμε μόνο εκτός, να κοιτάμε και μέσα τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί μόνο τότε θα είμαστε αξιόπιστοι προς τα έξω. Και επειδή δεν έχω χρόνο, θέλω να κάνω και έκκληση πράγματι να συνεχίσουμε με την αιρεσιμότητα, γιατί αλλιώς πάλι θα είμαστε στα προβλήματα. Καμπρίλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρία Είπατε, πρόσωπε. Σας ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για τον τρόπο με τον οποίο κάνατε τις διαβουλεύσεις. Οι ιδιαίτεροι μας έχουν εκφράσει ικανοποίηση. Είναι ένα θετικό σημείο κίνηση. Συγχαρητήρια επίση και για την αλλαγή τη προσέγγιση. Λιγότερε προτεραιότητε, περισσότερη αποτελεσματικότητα, περισσότερη ευελιξία. Θέλω να επιμείνω σε τρει πτυχέ. Πρώτον, χαιρόμαστε που τονίζετε το θέμα της μετανάστευσης και της ασφάλειας τι γίνεται με κοινή βάση δεδομένων στην οποία θα έχουν όλοι πρόσβαση για να αποφύγουμε την ε, λαθροδιακίνηση και την παρανομία. Πώς θα μπορέσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί δεν πρέπει να δώσουμε περισσότερη σημασία σε μια τέτοια βάση δεδομένων, χωρίς να αναμειγνιόμαστε στα εσωτερικά των γειτόνων μας, πρέπει να υπογραμμίσουμε το θέμα της εκπαίδευσης, γιατί αυτό μας εξυπηρετεί και εμάς. Και πώς θα προωθήσουμε την προβολή της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός πρέπει να είναι ένας στόχος μας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας. Ευχαριστώ. Πολύ κυρία Γκόμες. Συμφωνώ με τα όσα λέτε για τις οικονομικές εξελίξεις όσον αφορά την απασχόληση των νέων, αλλά είναι σημαντικό να πείσουμε και τις χώρες ε, μέλη να σταματήσουμε με αυτήν τη λιτότητα η οποία δημιουργεί σε περισσότερη ανεργία, σε περισσότερη αποξένωση των νέων και βέβαια στην αστικοποίηση των μεταναστών. Θα αρχίσουμε να συντονίζουμε τη δράση μας. Τώρα μάλιστα που θέλετε να συνδυάσετε αυτή την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονία με το άρθρο 42.7 και τις επιθέσεις στη Μέση Ανατολή, πώς θα τα συνδυάσετε αυτά τα δύο, πώς θα τα συντονίσετε. Η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία, τι ρόλο παίζουν. Τι θα κάνουμε με αυτές, πώς θα αποφύγουμε και τους λαθροδιακινητές να συνεχίσουν τη δουλειά τους αν δεν ανοίξουμε ασφαλή σύνορα για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Γιατί αυτοί οι πρόσφυγες προσπαθούν να ξεφύγουν από αυτούς που οδήγησαν στις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι. Και όχι να τους εμποδίζουμε να έρθουν. Σταματήστε λέει ο πρόεδρος, έληξε ο χρόνος σας. Η κυρία Σχάκ έχει τώρα το λόγο. Πάντα είναι ένα καλό παράδειγμα γιατί τελεί το χρόνο τη. Ευχαριστώ, είπατε εκπρόσωπε Επιτροπε Χάνε, ευχαριστώ που ήρθατε να μας ε, μιλήσετε σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς με τόσο περιορισμένο χρόνο. Σας ευχαριστούμε για το εγγραφό σας. Είναι αποτελεί καλή βάση και μπορεί να μας βοηθήσει να δώσουμε νόημα στη σχέση μας με τις γείτονες χώρες. Στην πράξη όμως πώς θα γίνουν αυτά, γιατί όταν υποσχόμεθα περισσότερα και περισσότερα δεν το κάνουμε συχνά και δεν ακολουθούμε το πνεύμα επαρκώς. Η αστάθεια σημαίνει τελικά σχέσεις από κυβέρνηση με κυβέρνηση, ενώ οι ίδιες κυβερνήσεις είναι αυτές που καταπιέζουν τον πληθυσμό τους και κυρίως τους νέους. Μακροπρόθεσμα λοιπόν, αν δεν δώσουμε περισσότερο νόημα για περισσότερη απασχόληση σε αυτούς τους νέους ολόκληρη την Ευρώπη, θα οδηγηθούμε σε μια χαμένη γενιά που θα μας έρθει μπούμεραγκ. Κυρίως λοιπόν αυτούς τους καιρούς που χρειαζόμαστε δράσεις αντιτομοκρατίας και ασφάλειας να διδαχτούμε από το παρελθόν και να μην κάνουμε τα ίδια σφάλματα. Να μην νομίζουμε ότι υπάρχει σταθερότητα και αυτή να υπάρχει μόνο στα λόγια ή να υπάρχει καταπιέζοντας όμως όλο και περισσότερο τον κόσμο. Πώς θα τα αναλύσετε όλα αυτά και στην πράξη πώς θα τα υλοποιήσετε. Ναι, καλό παράδειγμα, λέει ο πρόεδρο. Στηρίζετε το χρόνο σα. Ο κύριο Κέλλερ. Ευχαριστώ. Η πολιτική μα μέχρι τώρα ήταν να ενισχύσουμε την ασφάλειά μα, κυρίω στα εξωτερικά μα σύνορα. Η ερώτησή μου είναι η εξή. Οι δηλώσει μα, τα σχέδιά μα συνοδεύονται από την κατάλληλη χρηματοδότηση. Έχω υπόψη μου την εσωτερική ασφάλεια και τη συμφωνία για τα στοιχεία επιβατών ε, αεροπορικών ε, εταιριών. Είναι πράγματα και στοιχεία το οποίο η έχει πει ότι τα θέλει. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάποια στρατηγική για τη Μέση Ανατολή. Για το Κουρδιστάν, για παράδειγμα. Άκουσα ότι ο κύριος Πούτιν υποσχέθηκε αναγνώριση. Ποια είναι η αντίδρασή σας. Τρίτον, πρέπει να διαλέξουμε ανάμεσα σε δύο κακά. Τα σχέδια του κύριου Πούτιν θα μας οδηγήσουν στο σενάριο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος που λειτουργήσε αλλά είχε κάποιο τίμημα. Κόβεται το μικρόφωνο του μιλητή. Κυρία Γκίλ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, είπατε εκπρόσωπε, κύριε Επίτροπε, έχουμε μια στρατηγική γειτονία εδώ και δύο δεκαετίες και έχουμε αφιερώσει αρκετούς πόρους. Η γειτονιά μας λοιπόν είναι σε αναταραχή και πράγματι δεν υπάρχει οικονομική ευημερία και αναγνωρίζω ποιο, πώς η στρατηγική αυτή έχει υπονομευθεί από τα κράτη-μέλη που το καθένα ακολουθεί το δικό του πρόγραμμα. Το θέμα είναι λοιπόν πώς θα έχουμε περισσότερη αποτελεσματικότητα. Είπατε πως συναντηθήκατε με τους πρέσβεις των χωρών εταίρων από τα κράτη-μέλη είχατε κάποια συνεισφορά. Δεύτερον, υπάρχουν πολλές ε, ανησυχίες ασφαλείας μετά την ε, επίθεση, τις επιθέσεις στο Παρίσι για την ευκολία με την οποία βρίσκουμε Καλάσνικοφ ε, και στις γειτονικέ χώρες και ξέρω πως οι χώρες εταίροι αρνούνται να κάνουν κάτι. Τι σκοπεύετε να κάνετε γι' αυτό. Σας ευχαριστώ. Κύριε Κούζο το, το μικρόφωνο του ομιλητή. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρία Μογκερίνη, κύριε Επίτροπε. Η πολιτική αυτή γειτονία και η ανθεώρησή τη θα αποτύχει και πάλι, γιατί για μένα δεν χρησιμοποιεί μια συμμετρία οικονομική ή άλλη. Προσπαθούμε να βρούμε αντί για εταίρους υποτακτικούς. Πώς θα λύσουμε τις ε, παγωμένες συγκρούσεις, είτε πρόκειται για την Παλαιστίνη, είτε για την Κύπρο, είτε για την ε, Σαχάρα. Γιατί κάνουμε παρεμβάσεις και δεν κοιτάμε πώς φτάνουν τα όπλα. Το 42-7 σημαίνει στρατικοποίηση της Ευρώπης. Υπάρχει ασυμμετρική απειλή. Σαχέλ και αλλού γίνονται λαθρεμπόριο πετρελαίου. Και αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ. Τελευταίο ο κ. Σπανιό. Euh, το είπατε και η πολιτική γειτονία πρέπει να αλλάξει. Φτάσαμε στα όρια τη προηγούμενη πολιτική μα τώρα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι και το ξέρουμε. Το 2015 δεν έχει καμία σύγκριση με το 2003. Πρώτη παρατήρηση. Πώ μπορεί η πολιτική μα να διευκολύνει την σταθεροποίηση στι χώρε τη γειτονία διότι η περισσότερη Ευρώπη είναι κάτι που ικανοποιεί τους εθνικιστές και τους αντιευρωπαϊστές. Επίσης, ε, η πολιτική γειτονία δεν απαιτεί να συνεργαστούμε με, τους, με τις χώρες εταίρους, όμως δεν μπορούμε να σκεφτούμε την νότια όχθη της Μεσογείου χωρίς τους μεγάλους πρωταγωνιστές της Μέσης Ανατολής. Πώ μπορούμε λοιπόν όλα αυτά να είναι αρμονικά, δεν πρέπει να υπάρχει συστηματική συνεργασία με τον Αραβικό Σύνδεσμο και τι χώρε του. Θα πρέπει επίσης να σκεφτούμε την Σύνοδο Αφρικής Ευρώπης ε, και εκεί να σκεφτούμε τον καθοριστικό ρόλο της Μεσογείου. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για να αποφύγουμε την ρίζοσπαστικοποίηση των γειτόνων μας. Σας ευχαριστώ για τη συζήτηση. Είναι νομίζω σημαντικό στην ε, έκθεση προόδου να αφιερώσουμε μια μέρα ίσως σε κάθε χώρα γιατί υπάρχουν πολλές διαφορές αλλά βεβαίως ε, από την άλλη λέμε πως είναι μία και ενιαία η στρατηγική. Υπάρχει λοιπόν μία αντίφαση εδώ πέρα οπότε δεν ξέρω το αυτό το ότι κάνουμε χωριστές εκθέσεις ε, για την κάθε χώρα πως οδηγεί στο να χάνουμε την ενιαία στρατηγική. Κυρία Μογκερίνη, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Η αναθεώρηση τη Ευρωπαϊκή Πολιτική γειτονία είναι μέρο τη εξωτερική μα πολιτική. Κάποιοι από εσά το είπατε ότι περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων εγχειρημάτων. Πρόκειται για ένα στοιχείο κλειδί που όμως δεν ικανοποιεί τα πάντα και δεν αφορά τα πάντα. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα κυρίως η διαδικασία μέσα στην οποία βρισκόμαστε με τους εταίρους μας, γιατί έτσι κατανοούμε καλύτερα τους εταίρους μας και βάζουμε τις βάσεις για πιο αποτελεσματική συνεργασία. Αλλά αν πιστεύετε ότι αυτό θα λύσει όλα τα προβλήματα, από το κουρδικό μέχρι το κυπριακό και την Μέση Ανατολή, υπάρχουν και άλλα μέσα. Πολύ σημαντικό λοιπόν, αλλά να ξέρουμε ποιο είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο βρίσκεται. Επειδή το Μποργέτσιο δεν είναι εδώ πια, λυπάμαι, αλλά εκείνος είπε να μην συνεχίσουμε να κάνουμε business as usual, ίσως γι' αυτό δεν βρίσκεται και αυτός εδώ πια και γι' αυτό έφυγε, αλλά πιστέψτε με, τίποτα από αυτά που κάνουμε αυτό το χρόνο που έχουμε αναλάβει τα καθήκοντά μας δεν είναι business as usual. Σήμερα το πρωί αρχίσαμε λέγοντας ότι ίσω είναι η τελευταία ευκαιρία, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια νέα αρχή. Ήταν η πρώτη φορά που είχαμε μια τέτοια διαχείριση κρίσης. Δεν ήταν μάλλον η πρώτη φορά που είχαμε διαχείριση κρίση από τότε που αναλάβαμε τα καθήκοντά μα. Για μα το business as usual είναι η επίλυση των κρίσεων, γιατί συνεχώ τι έχουμε. Πριν από ένα μήνα Όλοι λέγατε μετανάστευση, μετανάστευση, μετανάστευση. Σήμερα λέτε τρομοκρατία, τρομοκρατία, τρομοκρατία. Όλα αυτά πρέπει να τα κρατήσουμε, να τα ασχοληθούμε και ευχαριστώ που κάποιος μίλησε και για νέες ευκαιρίες που έχουμε μπροστά μας. Είναι αλήθεια ότι η εταιρική σχέση έχει περισσότερη σημασία τώρα από ό,τι είχε το 2003. Γιατί έχουμε κοινού κινδύνους και κοινέ ευκαιρίες μαζί. Άρα διαχείριση κρίσεων είναι επίσης ένα κοινό μας καθήκον και συνεχείς επενδύσεις. Τώρα είναι σαφές ότι η ασφάλεια απαιτεί συνεργασία και κάποιες επιλογές ΚΕΠΑ. Είναι κάτι που και αυτό πρέπει να μπει στην όλη εικόνα, ξέροντας τι ισχύει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τι εκτός. Και η μετανάστευση είναι το δεύτερο σκέλος. Τώρα κάποιοι από εσά αναφερθήκατε στην παράτυπη μετανάστευση από τις γείτονες χώρες. Δείτε τα νούμερα. Οι πρόσφυγες που έρχονται εδώ δεν έρχονται από τις χώρες της ε, νότιας γειτονίας, έρχονται μέσω αυτών ίσως και οι ίδιες οι χώρες της νότιας γειτονίας μας έχουν κατακλειστεί από πρόσφυγες. Είμαστε στην ίδια πλευρά με αυτούς, προσπαθούμε μαζί τους να διαχειριστούμε το πρόβλημα. Υπάρχει μια αλλαγή που ίσως ε, αργούμε ως Ευρωπαίοι να αντιληφθούμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι με τους νότιους γείτονές μας βρισκόμαστε από την ίδια μεριά του προβλήματος. Τώρα για τις αραβικές χώρες. Έχουμε κοινέ υπουργικέ συναντήσεις, τακτικά και κάποιες διασκέψεις όπου προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και αυτοί έχουν τα δικά τους εσωτερικά προβλήματα να λύσουν. Το πραγματικό πάντως πρόβλημα για μένα είναι ακριβώς αυτή η χαμένη γενιά. Γι' αυτό και μίλησα για οικονομικές ευκαιρίες που πρέπει να δώσουμε και να προσφέρουμε. Ξεχνάμε ήδη την Αραβική Άνοιξη. Το πραγματικό όμως ζήτημα είναι το δημογραφικό. Η οικονομία και το γεγονός ότι έχουμε τόσο πολλούς νέους με προσόντα που έχουν εκπαίδευση που όχι μόνο βρίσκονται στην ανεργία μερικές φορές είναι αυτοί που μας απειλούν. Αυτό είναι κάτι που ισχύει σε όλες τις χώρες γειτονίας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια. Αυτό λοιπόν είναι το στοιχείο κλειδί. Το περισσότερα για περισσότερα και λιγότερα για λιγότερα το αφήνω για τον Επίτροπο Χάν. Πάντως, το ζήτημα είναι ότι πρέπει να βρούμε τρόπους με τους εταίρους μας. Και οι εταίροι μας δεν είναι μόνο οι κυβερνήσεις, είναι ο κόσμος. Όπως εμείς δεν είμαστε μόνο οι θεσμοί, είμαστε και ο λαός της Ευρώπης. Πρέπει λοιπόν να βρούμε τρόπους να ε, φτιάξουμε οι κοινωνίες οι οποίες να αντιστέκονται καλύτερα, στις οποίες να συμμετέχουν όλοι και που να είναι ασφαλείς. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος και σταθερές. Ο μόνος τρόπος για να πετύχουμε την ασφάλεια είναι ισχυρά ανθρώπινα δικαιώματα και συμμετοχή όλων. Δεν είναι σε αντίθεση αυτά μεταξύ τους. Για το 42-7 είμαι έτοιμη να σας δώσω ότι σημειώματα υπάρχουν. Ευχαρίστως. Τις τελευταίες 48 ώρες έτσι και αλλιώς δουλεύουμε σκληρά πάνω σε αυτό. Είναι η πρώτη φορά που ενεργοποιείται αυτό το άρθρο, οπότε χρειαζόταν σκληρή προετοιμασία από την πλευρά μας. Ευχαρίστως λοιπόν μοιραστώ μαζί σας ότι έχουμε και να συνεργαστούμε. Και εγώ, όποτε είμαι στις Βρυξέλλες, ευχαρίστως μεταξύ μας, σε περιορισμένο κύκλο, να συζητούμε περισσότερες λεπτομέρειες. Ευχαριστώ. Πρόεδρος εκτός μικροφώνου. Κύριε κύριος Μποργέτσιο ζήτησε συγγνώμη είδατε πως είχε τα γελιά ηλίου λόγω της αρρώστιας και ε, πρέπει να πάει στο νοσοκομείο μου είπαν τώρα. Αυτά λοιπόν σας ε, ευχαριστώ για την προσφορά για το 42.7. Ε, από ό,τι κατάλαβα, Φεντερίκα, εσύ είσαι υπεύθυνη για το More ε, for More και ο Ιωάννης για το Less for Less, έτσι πάει. Ιωάννης έχετε το λόγο. Ναι, ναι, τα έχουμε μοιράσει καλά. Να σας διαβεβαιώσω πως δεν υπάρχει ε, ουσιαστική διαφοροποίηση μεταξύ Ανατολής ε, και Νότου. Έχουμε τα τμήματά μας, το προσωπικό μας, ε, είμαστε υποχρεωμένοι να συνεργαζόμαστε με τις διάφορες χώρες αλλά βεβαίως κάποια στιγμή δίνουμε περισσότερο βάρος σε μία ή την άλλη χώρα αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να υπάρξει μία ισότιμη αντιμετώπιση και των δύο περιοχών μια περισσότερη εξορροπιστεύσεων για το more for more. και εδώ πέρα θα πρέπει να υπάρξει μια λογική, λογικότερη εξέλιξη, να μην βλέπουμε τα πράγματα τόσο μηχανιστικά, αλλά να βλέπουμε ως μέτρο σύγκρισης και τις εσωτερικές εξελίξεις μιας ε, χώρας και όχι αυτά τα οποία έχουν εφαρμοστεί ως προδιαγραφές. Δηλαδή πρέπει να βοηθήσουμε τις ε, χώρες και το less for less, το λιγότερα για λιγότερα. Ε, κοιτάξτε, αυτό φαίνεται από το ότι παραδείγματο χάρη διαθέτουμε λιγότερα κονδύλια όταν απορροφούνται λιγότερα κονδύλια. Αλλά συνήθως αυτό έχει τη μορφή του ότι επενδύουμε στην κοινωνία των πολιτών η οποία σε πολλές από αυτές τις χώρες έχει μια σημαντική λειτουργία και την ενισχύουμε για να αναπτυχθεί. Αλλά εδώ πέρα βλέπουμε μια εξέλιξη που είναι δηλαδή ότι κάποιες χώρες ακολουθούν ε, το παράδειγμα της Ρωσίας και εμποδίζουν τη χρηματοδότηση μικιό από το εξωτερικό. Οπότε θα πρέπει να είμαστε κάποιο πιο ευέλικτοι και ρεαλιστικοί. Γενικά μπορώ να πω το εξή αυτό το οποίο είπε και είπα τι εκπρόσωπος. Δηλαδή θα πρέπει να δούμε και να αντιμετωπίσουμε και να αντιδρούμε ξεχωριστά σε κάθε χώρα για να, να βοηθήσουμε την οικονομική ανάπτυξη αλλά αυτό δεν σημαίνει μονοδιάστατα να επενδύσουμε στην οικονομία μιας χώρας αλλά να δημιουργούνται και θέσεις εργασίας ε, θέσεις μαθητείας ε, εκπαίδευσης όχι μόνο ακαδημαϊκής εκπαίδευσης αλλά και επαγγελματικής και αυτή ακριβώς είναι η ανησυχία κάποιων ε, χωρών γειτονικών στην οποία πρέπει να αντιδράσουμε δηλαδή να μην δημιουργήσουμε ένα φαινόμενο κεντρομόλο δηλαδή καλά εκπαιδευμένοι άνθρωποι ε, να φεύγουν ε, και να έρχονται στην Ευρώπη και να μένουν αυτές οι χώρες μετά πάλι στην ίδια κατάσταση να υπάρχει μια κυκλοφορία των ε, εγκεφάλων ε, αμφίδρομη. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να δημιουργήσουμε και προγράμματα χρηματοδότησης ε, των νέων επιχειρήσεων να εστιαστούμε στους νέους και όχι μόνο. Υπάρχει η δυνατότητα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότηση και ανάπτυξη και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να δημιουργήσουμε περισσότερη μόχλευση και να υποστηρίσουμε τις μικρόμεσες επιχειρήσεις. Οπότε εδώ πέρα δεν υπάρχουν όρια στην φαντασία θα έλεγε κανείς και τέλος πρέπει να συνεργαστούμε και με τον Αραβικό Σύνδεσμο. Είναι σημαντικό λοιπόν κάποιοι οργανισμοί εδώ πέρα να αναλάβουν κάποια καθήκοντα στον τομέα της αρμοδιότητάς τους γιατί είναι σημαντικοί συνομιλητέ για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πάλι λοιπόν σας ευχαριστώ για τη συνεργασία σας τους τελευταίους μήνες και όπως είπαμε τώρα ξεκινάει η ε, δουλειά. Ξέρετε πως τα χαρτιά είναι κάτι, αλλά είναι κάτι διαφορετικό η εφαρμογή. Σας ευχαριστώ κυρία Μογκερίνη, κύριε Χάν για αυτά τα οποία μας είπατε και σα ευχαριστώ που ήρθατε εδώ πριν από την συνέντευξη τύπου στην οποία σας εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ.